Ξέρετε ότι έχουμε το θέμα της ε, Ελβετίας, την απόφαση της Ελβετίας και θα ήθελα να ζητήσω μετά από την κυρία Πάκ να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης στη Βοσνία Ζεγοβίνη, η οποία είναι έκρηθμη. Υπάρχει Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία και μετά θα συνεχίσουμε με την φυσιολογική ημερήσια διάταξη. Για τα πρακτικά θα ακολουθήσουμε τη συνηθισμένη διαδικασία. Ελβετία. Εγώ δεν ξέρω αν έγινε και σε, στις χώρες σας, αλλά από χθες το βράδυ όλοι ζητούν συνέντευξη και ζητούν να με ρωτήσουν ποια θα έχουν δημιουργήσει μια κάποια αναστάτωση ήταν πολύ μικρή η πλειοψηφία και όπως φαίνεται στο γερμανόφωνο τμήμα υποστηρίχθηκε το δημοψήφισμα αυτό, όχι στο γαλλόφωνο, ακριβώς στο τμήμα αυτό το οποίο έχει τους λιγότερους ξένους όμως. Τα κρατήρια λοιπόν, τα καντόνια, τα ε, γερμανόφωνα υποστήριξαν αυτό το δημοψήφισμα. Όχι όμως το Τεστίνο. Υπάρχουν και οι, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται στην περιοχή του Τεσίνο και οι οποίοι παίζουν μεγάλο ρόλο στην τοπική οικονομία. Η άποψή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θα ήθελα να ακούσω την άποψη της ε, Επιτροπής μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα λόγο να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Οι συνθήκες ισχύουν, οι συμφωνίες ισχύουν. Πρέπει μέσα σε τρία χρόνια η ελβετική κυβέρνηση να κάνει μια πρόταση τροποποίησης των συμπεφωνημένων και τότε φυσικά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, θα, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προφανώς δεν μπορεί να είναι η Ελβετία μέσα στην ενιαία αγορά όταν η ελεύθερη κυκλοφορία δεν ισχύει για τους εργαζόμενους και για τα κεφάλαια στην Ελβετία. Αυτό ίσως είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα, αν θυγεί η ελευθερία διακίνηση των κεφαλαίων, λέει ο κύριος Μπρόκ. Αλλά φυσικά θα υπάρξουν και προβλήματα με τη, στη Γερμανία για τα θέματα συνεργασίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δεν υπάρχει λόγος να αναστατωθούμε. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις επαφές με τους Ελβετούς συναδέλφους μας. Ήταν προηγουμένως, πριν από δύο εβδομάδες, ε, η αντιπροσωπεία του Ελβετικού Κοινοβουλίου μέσα στους οποίους ήταν και κάποιος εκπρόσωπος του κόμματος που ζήτησε το δημοψήφισμα αυτό. Και θα πρέπει όμως να καταλάβουν οι Ελβετοί ότι δεν μπορούν επιλεκτικά να κάνουν συμφωνίες. Θα πρέπει, αν θέλουν να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζουν τις τέσσερις ελευθερίες οι οποίες ισχύουν βάσει της συνθήκης Λισαβόνας. Και δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν διμερείς μονάχα συμφωνίες με μεμονωμένες χώρες. Θα πρέπει να τηρήσουν την, ε, τις συμφωνίες αυτές και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι και αυτά τα οποία ζητά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πάντα και αυτά συνάδοντα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τίθεται και το θέμα της ε, ελευθερίας διακίνησης των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ε, και ένα ψήφισμα που θέλησαμε να διατυπώσουμε είναι πάρα πολύ σημαντική η ελευθερία διακίνησης, αλλά πάντα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης οι προβληματικές περιπτώσεις που σε επίπεδο ποσοστιαίο δεν είναι ουσιαστικές. Το ουσιαστικό είναι να εξασφαλίσουμε να μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας ότι η οποιαδήποτε κατάχρηση που γίνεται αυτού του, δια, του δικαιώματος είναι πάρα πολύ περιορισμένη και όχι να, βάλουμε, να βοηθήσουμε τους ε, αντιευρωπαϊστές να ενισχύσουν τη θέση τους. Σίγουρα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα εν καιρό της Ελβετίας. Έχετε εδώ κάποια ερωτήματα? Όχι. Κυρία Μουνίχ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή όταν το άξονα μου ήταν αστείο αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι είναι σοβαρό. Μπορεί κανείς να μιλήσει για την ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων, αλλά για τις τέσσερις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένοι θέλουν να τις θέσουν αμφιβόλο όταν λέγοντας ότι υπάρχουν καταχρήσεις. Αλλά οι καταχρήσεις δεν είναι επαρκείς για να λύσουν μια ελευθερία. Τα θέματα των διμερών συμφωνιών μας έχουν να κάνουν με τα το τραπεζικό απόρριτο, με τις μεταφορές, με πάρα πολλές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τμήμα της εσωτερικής αγοράς μας. Δηλαδή, εκτός που δεν είναι χώρα μέλος η Ελβετία, συμμετέχει σε όλες αυτές τις πολιτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε όμως και όχι να περιμένουμε μέσα σε τρία χρόνια να γίνει κάτι, ενώ η Ελβετία θα κάνει τα απαραίτητα για να εφαρμόσει τα αποτελέσματα αυτού του δημοψηφίσματος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν λανθασμένο να υπάρξει κάποιο υπόμνημα, κάποια δήλωση από την πλευρά της Επιτροπής μας. Παρακαλώ να με ακούσετε. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια δήλωση, ένα υπόμνημα της Επιτροπής μας, τονίζοντας ποιο είναι το πλαίσιο των σχέσεων μας με την Ελβετία, η οποία είναι μια τρίτη χώρα και η οποία δεν μπορεί να θέσει να αμφιβόλο τις βασικές αρχές που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων να πω ότι πραγματικά λυπούμεθα για αυτή την έκβαση του δημοψηφίσματος και ενδεχομένως ε, να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους των ε, πολιτικών να εκπονήσουν κάποιο υπόμνημα γιατί υπάρχουν και πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε, ας πούμε, ε, να γνωστοποιήσουν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις στα προγράμματα Εράσμους, όπως έμαθα ε, πρόσφατα, αλλά και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Καλό θα ήταν λοιπόν να καταγράψουμε τον αντίκτυπο ε, αυτών των αποφάσεων και βεβαίως να υποβάλουμε τα ζητήματα αυτά στους ελβετούς συνομιλητές μας. Κύριε Πρόεδρε, σας υποστηρίζω ανεπιφύλακτα και πράγματι δεν πρέπει τώρα να αντιδράσουμε παρορμητικά. Πρέπει να επιληφθούμε σοβαρά του θέματος και εγώ Πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με παραβίαση των συνθήκων και του ευρωπαϊκού δικαίου και δεν επιτρέπεται να κάνουμε καμία παραχώρηση. Όμως ε, πρέπει να γνωρίζουμε, η απόφαση είναι ότι ο νομοθέτης στην Ελβετία τα επόμενα τρία χρόνια οφείλει να καταθέσει νομοθετική πρόταση. Πρέπει λοιπόν στο νομοθέτη της ε, Ελβετίας ε, να του δημιουργήσουμε την πίεση να καταθέσει μια τέτοια πρόταση πρόταση η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και θα διαχωρίζει όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα υπόλοιπα. Αν όμως τώρα επιτεθούμε βεβαιασμένα, απλά το μόνο που θα κάνουμε είναι θα δώσουμε αέρα στα πανιά των λαϊκίστικων αντιδημοκρατικών δυνάμεων που θα πούνε ότι μόλις αποφανθεί ο λαός αυτομάτως επιβάλλονται κυρώσεις. Γιατί κάποιος μίλησε για το πρόγραμμα Έρασμος. Δεν πρέπει να προκαλέσουμε την εντύπωση ότι η δική μας απάντηση είναι πάρα αυτά κυρώσεις. Σαφώς και είμαι υπέρ μια σκληρής γραμμής, μην αμφιβάλλετε από αυτού, αλλά αυτή η σκληρή γραμμή θα πρέπει να βασίζεται σε αδιάσυστα γεγονότα. Και δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια στα χέρια μας μετά το χθεσινό ψήφισμα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα προτείνει η Ελβετία. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα πρέπει να καταλάβουν οι ότι η Ελβετία είναι η δημοκρατία και ε, αποφάσισε με τρόπο που ενδεχομένως δεν τους πολύ αρέσει, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να τους πούμε θα ψηφίσετε και θα ξαναψηφίσετε μέχρι το αποτέλεσμα να ικανοποιεί εμάς. Είναι γεγονός ότι με τις δημοκρατικές τους διαδικασίες ψήφισαν και αποφάσισαν. Και η έκβαση μπορεί να μην μας ικανοποιεί, αλλά έχουν απόλυτο δικαίωμα να αποφασίσουν όπως θέλουν. Και θα, θα, θα συμφωνήσω με τον Μπέρν. Δεν είναι δυνατόν εμείς να αποφασίσουμε αμέσως να απαντήσουμε με αντικυρώσεις ή με κυρώσει γιατί κανείς θα μπορεί να πει ότι ακριβώς επειδή δεν συμφωνούν με κάποια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό ακριβώς πήραν αυτήν την ε, απόφαση. Ε, φαντάζομαι ότι ε, εάν ε, τέτοια δημοψηφίσματα γίνονται και σε άλλες χώρες και στη δικιά σας πρόεδρε και στη δικιά μου, ίσως τα αποτελέσματα να ήταν παρόμοια. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να υπερβούμε το εμπόδιο αυτό, αυτή τη δυσκολία με ευφυΐα, με εξυπνάδα και όχι να δημιουργήσουμε προβλήματα περισσότερα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι και στην Ελβετία υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν τρομάξει με το αποτέλεσμα, κυρίως οι επιστήμονες, οι ερευνητές. Ε, στο ραδιόφωνο μόλις τώρα άκουσα έναν καθηγητή που είπε ότι το κύρος μας ε, ως ε, χώρα επιστήμης και έρευνας ε, θα καταστραφεί και θα καταστρέφεται αν δεν είχαμε αυτούς που έχουμε εδώ, Γερμανούς, Γάλλους, 31-20% αντίστοιχα, πολυδιδάσκουν, ερευνούν. Και όπως είπες και εσύ, αυτό το αποτέλεσμα, ε, η απόρριψη δηλαδή, προέρχεται κυρίως από τις γερμανόφωνες περιοχές και τώρα πολλοί το εκμεταλλεύονται για πολιτικούς ίδιους ε, σκοπούς. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πράγματι δεν πρέπει να βιαστούμε, αλλά να τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε. Ε, εντάξει, μπορείτε να αποφασίσετε διαφορετικά. Αν όμως συμβεί αυτό, τότε και εμείς θα δώσουμε μία απάντηση. Αλλά δεν θα πρέπει μετά από πόνερα να πετάξουμε και το μωρό, να περιμένουμε λιγάκι. Εγώ θέλω να πω κάτι μετά από αυτά ε, που είδα εχθέ στην τηλεόραση και εγώ ήμουν εκεί και η γυναίκα μου είπε ότι τη άρεσε πολύ το φουλάρι που φόραγα. Τώρα, αν πήγαινε με το σακάκι, από αυτού μπορούμε να τσακωθούμε. τα αφήνω αυτά τώρα. Όπω είπε και στην άλλη, δεν πρέπει με τα πόνερα να πετάξουμε και το μωρό. Να δούμε λιγάκι τι έγινε. Ε, ψήφισαν. Ε, 19.500 άνθρωποι και οι οικονομικές επιτυχίες ε, δεν προβλήθηκαν. Έχουμε ανθρώπους ε, με πολύ ψηλούς μισθούς, ε, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι εκδιώκουν τους άλλους. Νομίζω ότι όλα αυτά ε, έγιναν σε κύκλους όπου περνάει ο λαϊκισμός. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί και έχουμε βέβαια τρία χρόνια στη διάθεσή, μου, στη διάθεσή μας να δούμε τα κάνουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας θα κάνει μια περιήγηση, θα ξεκινήσει από το Βερολίνο και μπορούμε πάρα πολλά να τα συζητήσουμε. Ε, να πούμε ξεκάθαρα ξεκάθαρα τι ακριβώς ε, σημαίνουν οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τα επτά κεφάλαια. Αυτό που με ανησυχεί είναι αυτός από την Αυστρία, ε, του ΕΦΕ και η Μαρίν Λεπέν και οι ε, Βρετανοί και ο Φάρατς να του πούμε ότι είναι σπίτι σου, δεν σε θέλουμε εδώ. Ε, όταν λοιπόν ε, μιλάει ένας ε, πρωθυπουργός, ο ε, μιλάει και γελάει ειρωνικά, αυτό με ενοχλεί πολύ περισσότερο από αυτό που αποφάσισαν οι Ελβετοί. Δικαίωμά τους είναι, δεν τίθεται θέμα επ' αυτού και ένα θέμα να είναι σαφές και σε εμά υπάρχουν πολλοί λαϊκιστές, που το φθινόπωρο λένε το α και το Χριστούγεννα κάτι τελείως διαφορετικό. Μόνο που το να ε, χαράσει κανείς πολιτική με αυτά που ε, κατά καιρού λέγονται, αυτό δεν είναι σωστό. Να παραμείνουμε νυφάλοι, να μην αποφασίσουμε ε, πάρα αυτά κυρώσεις και νομίζω ότι θα ήταν και καλό να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις αποφάσεις ε, του λαού και κυρίως όχι των ορεινών, ε, των κατοίκων σε ορεινές περιοχές γιατί και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα ήθελα ε, να σας αντιπαραθέσω εδώ ε, το παράδειγμα της Βαβαρίας και τι έγινε στη Βαυαρία. Αλλά εντάξει, ας το αφήσω καλύτερα προς το παρόν. Ο κύριος Χάουιτ. Δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κάνουμε συζήτηση για τα θέματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που θέσατε αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρο. Εγώ συμφωνώ με τον Βρετανό συντηρητικό συνάδελφό μου ότι το να έχουμε μια απειλητική γλώσσα αυτό είναι αντιπαραγωγικό και θα πρέπει να έχουμε μια ήπια αντιμετώπιση για μια χώρα όπως η Ελβετία. Αλλά πιστεύω ότι είναι απόλυτα σαφές το ότι μπορούμε να πούμε, είναι σωστό να πούμε ότι υπάρχουν σουν ότι πρέπει να τηρούνται διεθνείς υποχρεώσεις και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει και το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί υπάρχουν πολλοί στη χώρα μου οι οποίοι θέλουν να τηρηθούν οι συνθήκες και δεν τις διαμφισβητούν θέλουν να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γενικά για το καλό όλων των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν βλέπουν ότι μια ε, διαφορετική μεταχείριση για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο σωστός δρόμος για το μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αναφερθούν και στην Επιτροπή μας και πιστεύω ότι είναι απόλυτα δημοκρατικό το να γίνεται ένα δημοψήφισμα και να αντλούνται συμπεράσματα από τη θέληση της πλειοψηφίας. Αυτό δεν πρέπει να το κρίνουμε εμεί το αποτέλεσμα. Αλλά τη στιγμή που υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες που επιβάλλουν υποχρεώσεις και όχι μονάχα δικαιώματα, είναι σαφές ότι αν δεν τηρεί κανείς τα καθήκοντά του, τις υποχρεώσεις του, δεν μπορεί να αναμένει να διατηρήσει και τα δικαιώματά του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στο διεθνή διπλωματικό στίβο και πρέπει να περιμένουμε όχι από μία ή δύο χώρες, αλλά από όλες τις χώρες μας μια αντίστοιχη στάση. Εντάξει, λέω ευχαριστώ. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να αναλύσουμε την ε, νομική κατάσταση. Βέβαια ε, θα πρέπει να ξέρει ότι αν κάποιος αρχίσει να ε, φεύγει από τους κανόνες, να βγαίνει από τη συνθήκη, αυτό μπορεί να οδηγήσει και άλλους. Υπάρχουν κάποιοι αυτοματισμοί οι οποίοι ίσως δεν πρέπει να ισχύουν πια. Θα πρέπει να αντλήσουμε ορισμένα συμπεράσματα από όλα αυτά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Συμβούλιο των Υπουργών με την Ομοφωνία. Ενδεχομένω θα είναι χρήσιμο να καλέσουμε και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, τον κύριο Σάλιβαν, να μα παρουσιάσει την άποψή του και να μα δώσει τι διευκρινήσει σε σχέση με το πώ βλέπει το Συμβούλιο την κατάσταση τη Ελβετία. Εγώ φυσικά δεν αμφισβητώ ότι είναι μια δημοκρατική απόφαση, αλλά υπάρχουν συνθήκε που συνδέουν με την, ε, την Ελβετία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί κανεί να ικανοποιεί ένα τμήμα των συνθήκων αυτών, αλλά όχι το υπόλοιπο. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι κάτι το εφικτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες ισχύουν. Όλα αυτά λοιπόν τα νομικά θέματα πρέπει να τα ελέγξουμε Σίλβιο είπε να μιλήσουμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ελβετίας και ίσως να περιμένουμε λιγάκι να δούμε ε, κατά πόσο τον ε, Μάρτιο ή τον Απρίλιο θα μπορούσαμε να φέρουμε κάτι στο Στρασβούργο, στην ε, Ολομέλεια και ενδεχομένω πριν από την επόμενη ε, συνάντησή μας μπορούμε να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να κάνει κανείς επί τη βάση των ε, νομικών ε, γνωμοδοτήσεων που θα πάρουμε και νομίζω ότι προς το παρόν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα εκεί που βρίσκονται, δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ε, θέλω λοιπόν να πω και στον κύριο Watson ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση και την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα είχε νόημα να μεταβούμε και στην ε, Ελβετία. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Η Ντόρις. Χωρίς μικρόφωνο η Ντόρις. Ήμουνα στη... στη Βοσνία στη... το Σαββατοκύριακο γιατί εκεί θα ξεκινούσε ένα χειμωνιάτικο φεστιβάλ. Δυστυχώς το μικρόφωνο της ομιλήτριας κάνει πολλά παράστα. <laughs> Does it work now? Yeah. Ich war am Freitag. Ήμουνα το, στο Σεράγεβο την Παρασκευή μαζί με διάφορους καλλιτεχνικούς δημιουργούς οι οποίοι θα ξεκινούσαν την εκδήλωση αυτού του καλλιτεχνικού φεστιβάλ που έχει κρατήσει εδώ και 35 χρόνια, ακόμα και την εποχή του πολέμου της Ιουκοσλαβίας, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε λόγω των διαδηλώσεων που στην αρχή ήταν ειρηνικέ. Θέλαμε λοιπόν να κηρύξουμε την έναρξη του φεστιβάλ, αλλά ήταν πολύ λίγοι οι οποίοι ήταν παρόντες, γιατί εμποδιστήκανε από τους διαδηλωτές, οι οποίοι ήταν 400 μέτρα πιο πέρα και είχαν κλείσει τον δρόμο. Θέλησαμε να πάμε στο θέατρο για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, αλλά είδαμε ότι αυτή η διαδήλωση δεν ήταν μονάχα ειρηνική πια, είχε και χούλιγανς οι οποίοι έβαλα φωτιά σε σπίτια, σε αυτοκίνητα της αστυνομία, σε γραφεία κυβερνητικά, υπήρξε μια κλιμάκωση εγώ πιστεύω ότι υπήρξε πραγματικά χειραγώγηση αυτής της διαδήλωσης από ορισμένους οι οποίοι κινούσαν τα νήματα και τους οποίους δεν μπορώ να κατονομάσω, δεν ξέρω ποιοι είναι. Αλλά το ίδιο έγινε και στην ε, Τούσλα όταν κατέβηκε στην αρχή της εβδομάδας κατέβηκαν 50.000 άτομα στους δρόμους. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ήταν εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν συγκεκριμένες διεκδικήσεις που θέλανε να φέρουν στην ε, δημοσιότητα γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εξουσία. Ξέρετε ότι η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι διαιρημένη σε δύο οντότητες. Η μία είναι Βοσνιακο-Κροατική Ομοσπονδία και περιλαμβάνει 10 καντόνια όπου έχουμε 10 πρωθυπουργού, έχουμε 10 κυβερνήσει που το καθένα κάνει περίπου ό,τι θέλει. Και αυτό δεν οδηγεί σε μεγάλη ικανοποίηση μεταξύ του πληθυσμού και αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η μεγάλη διαδήλωση στο Σεράγεβο, η οποία οδηγήθηκε σε μια σε μεγάλες διαδηλώσεις και το ίδιο έγινε στο Μόσταρ και σε άλλες πόλεις της περιοχής. Και στο Βοσνιακό λοιπόν και στο Κροατικό τμήμα της Βοσνιοκροαστικής Ομοσπονδίας υπήρξαν αυτές οι διαδηλώσεις που κατέληξαν σε βίες ενέργειες και εμπρισμούς. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι Ε, ικανοποιητική σε ένα καντόνι κοντά στο Μπίχατς. Ο πρωθυπουργός του καντονιού έτυχε επιθέσεως στο σπίτι του και έγιναν βλάβες στην οικία του. Εμείς που γνωρίζουμε πολύ καλά τη Βοσνία, ξέραμε ότι αυτό ήδη ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το προβλέψαμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δρούν ως χούλιγκαν στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Σε ορισμένε περιπτώσεις τώρα έχει υπάρξει και παρέτηση πρωθυπουργών από τρία καντόνια, αν θυμάμαι καλά. Και άλλοι έχουν πει ότι διαφωνούν τελείως με αυτά τα, τις διαδηλώσεις, αλλά υπάρχει μια γενική δυσφορία υπάρχουν εθνοτικά προβλήματα τα οποία οδηγούν στο να κατεβαίνει ο κόσμος και στο δρόμο και είναι αυτά που είπαμε και στην ε, έκθεση που ψηφίσαμε ως κοινοβούλιο πρόσφατα ότι οι επικεφαλής των κατονίων δεν συνεργάζονται καθόλου. Αυτό δεν τους βοηθάει να φέρει τη χώρα τους πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουν καθόλου να αντιμετωπίσουν τα καυτά προβλήματα της χώρας τους. και ελπίζω ότι θα μπορέσουν μετά από όλες αυτές τις καταστάσεις να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν με περισσότερη ελπίδα στους πολίτες τους και να προχωρήσουν προς μια κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να πει κανείς στους ηγέτες της Βοσνίας όχι μόνο εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όταν λέμε εμεί κάτι σε αυτού δεν μα ακούνε. Όταν το πει ο λαό όμω η Βοσνία Ερχοβίνη, τότε ίσω να αρχίσουν να καταλαβαίνουν οι ηγέτε. Από την άλλη πλευρά, στη Ρεπούμπλικα Σέρψκα υπήρξαν ε, κάποιες μικρές ε, διαδηλώσει, οι οποίες δεν οδήγησαν σε τίποτα αλλά ο πρόεδρος τη Ρεπούμπλικα Σέρψκα μαζί με τον Μπόζιτς, τον ηγέτη του ΕΣΔΕΣ, πήγε στο Βελιγράδι και είδανε τον κύριο Βούτσιτς και είναι γεγονός ότι αν ξεκινήσει τώρα μια τέτοια κατάσταση αυτή μπορεί να επεκταθεί σε όλη την χώρα, σε όλη τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Είναι πολλοί στην Βοσνία Ζεγοβίνη οι οποίοι ζητούν να προταχθούν οι εκλογές οι οποίες προβλέπονται για τον Οκτώβριο να γίνουν πιο, πιο νωρίς αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι εμείς δεν ξέρουμε ποιος κινεί τα νήματα. Τι ακριβώς θέλουν να επιδιώξουν και αν απλώς είναι μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν την ε, δυσφορία του κόμματος, αν υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα τα οποία υποκρύπτονται πίσω από όλα αυτά και αν τα πολιτικά κόμματα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ενέργειες αυτές και τον χουλιγανισμό για να περάσουν την δική τους θέση. Εγώ ίσως συνέβαλα όταν είπα ότι πρέπει να ξυπνήσουν πια οι πολίτες και να κάνουν κάτι για αυτή την κατάσταση. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί να παίξει και αυτό κάποιο ρόλο στην κατάσταση αυτή, αλλά πρέπει να είμαστε σόφρονες, να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Η Κομισιόν έχει δράσει πιστεύω με έναν τρόπο ο οποίος ήταν αρκετά σόφρον. Και η βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η δυσφορία του λαού γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνία, κανείς δεν ενδιαφέρεται για την καλύτερη οικονομική ανάπτυξη, για την καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση. Όλα αυτά γίνονται μεταξύ, μέσα σε εθνοτικά όρια και απλώς μοιράζονται τα χρήματα, υπάρχει απόλυτη δι, μόνιμη διαφθορά. Όταν μιλάει κανείς με τους ταξιτζίδες, όταν μιλάει κανείς με τον κόσμο στον δρόμο, το σύστημα είναι απόλυτα διεφθαρμένο και η πολιτική το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει να γεμίσουν τις τσέπες τους και όχι να βοηθήσουν τους πολίτες. Αυτά μας λένε οι πολίτες και επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με την εταιρικού χαρακτήρα συμφωνία με τη Βοσνία. Και αυτοί οι οποίοι θέλουν να κατέβουν και να διαδηλώσουν με αξιοπρέπεια, ακόμα και αυτοί θέλουν να τονίσουν ότι δεν υπάρχει χώρος για χουλικανισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλα αυτά που είπε η κυρία Πακ μόλις τώρα. Κυρίως δε για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός ανάμεσα σε μια κοινωνική εξέγερση, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από κοινωνικής απόψεως και το κομμάτι το οποίο το οποίο αφορά ε, την ε, ε, χειραγώγηση της κοινή γνώμης. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι όντως οι οποίοι θέλουν, επιδιώκουν μάλλον, πολιτικά ωφέλη από αυτήν την κατάσταση. Αυτό είναι επικίνδυνο. Η κατάσταση είναι επικίνδυνο. Στο Μοστάρα, ας πούμε, περνώντας από το ανατολικό στο δυτικό τμήμα, ε, με φωνάζοντας πολύ προκλητικά συνθήματα, αυτό ξεκινάει μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επομένως ε, και μπορεί να καταλήξει σε σύραξη μεταξύ των λαών, μεταξύ των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει τον ηγετικό της ε, ρόλο ε, και νομίζω ότι κατά αυτή την έννοια θα είναι και επικοδομητική η αυριανή συζήτηση με την ε, Κάθριν Άστον. Ε, πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη. Δεν θα πρέπει να ριζοσπαστικοποιηθεί περισσότερο και το μήνυμα θα πρέπει να είναι σαφές από την πλευρά. Ο εξτρεμισμός, η κάθε μορφή προσπάθεια ανεξαρτοποίησης κτλ. αποτελούν στην ουσία τροχοπέδι προς το μέλλον της Ευρωπαϊκής, ε, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Κύριε Πρόεδρε, Αυτά που είπε μόλις τώρα η κυρία Ντόρις Πακ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι θέλω να τα υποστηρίξω ανεπιφύλατα. Την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη στην Ολομέλεια, είπα ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει κάποια διαμαρτυρία. Αυτές οι διαμαρτυρίες όμως ε, εντωμεταξύ έχουν ξεπεραστεί. Ξεκίνησαν πριν από αρκετό καιρό ως ένα είδος εξέγερσης των νέων. Εντωμεταξύ όμως έχουν ε, εκτραχυνθεί και μέσα σε αυτές τις κινήσεις των φοιτητών έχουν παρισ Φρύση, χαοτική, χούλιγκανς και άλλοι. Αν δούμε λοιπόν τα αιτήματα, ε, μεταξύ άλλων θα διαπιστώσουμε ότι η SDA ζητάει πρόορες εκλογές, αλλά ξέρετε τι θα γίνει, θα εκλεγούν πάλι οι ίδιοι αυτοί που είναι σήμερα, ίσως με διαφορετική σύνθεση με άλλα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιληφθούμε πιο σοβαρά του θέματος. Έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική ε, τάξη που εξοργίζει τους πολίτες, όσοι δεν εξοργίζονται φεύγουν, γιατί φεύγουν πάρα πολύ από τη Βοσνία Ζεγοβίνη οι υπόλοιποι ρίζοσπαστικοποιούνται και εμείς, μην ξεχνάτε, δαπανάμε πάρα πολλά κονδύλια, έχουμε ε, δυνάμεις τις οποίες συντηρούμε στην ε, Βοσνία Ερσεγοβίνη. Είναι πολύ δαπανηρό και αυτό, αλλά δεν έχει συνεισφέρει πουθενά. Ε, πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας. Και μην ξεχνάμε ότι και εμείς φέρουμε ευθύνη, γιατί η συνθήκη του Ντέιτον και το κείμενο σύνταγμα, ναι μεν τότε έθεσαν τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν έφεραν τη λύση. Η πολιτική της Βοσνίας μόνοι τους και οι κινήσει διαμαρτυρίας μόνες τους δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι πρέπει επιγόντως να επιληφθεί του θέματος η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βοσνίας Αρσεγοβίνης γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα υπάρξει μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Πρόεδρος, Περνάμε τώρα στην κανονική ημερήσια διάταξη, αυτή που είχε προβλεφθεί. Πρόκειται για την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η συγκίτρια είναι η κυρία Μαρία Μουνίς Ντε Ουρκίζα. Μισό λεπτό όμως να μιλήσει κάποιος για την Βοσνία πριν περάσουμε στην απαλλαγή. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να στηρίξω την συνάδελφο Ντόρις Πάκα αλλά και ε, αυτά που είπε ο συνάδελφος Απόσελτ μόλις τώρα. Πραγματικά, ειλικρινά, θα ήθελα να σας ζητήσω να ενεργήσετε με τρόπο ώστε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη πού συμβαίνουν τα διάφορα, με ποιο τρόπο, ποιες είναι οι δυνάμεις ε, που εμπλέκονται. Να σας πω ότι χθες όλη τη μέρα παρακολουθούσα την ε, κατάσταση. Ε, διάβαζα, άκουγα τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα διάφορα πρακτορία και από την Κροατία, κροατικά μέσα αλλά και άλλα. Υπάρχουν πρόδρομα σημάδια και βέβαια εδώ δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, θα το καταλάβετε όλοι. Γιατί στην ουσία ε, ένας λαός έχει ε, εξηγερθεί στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Στο Μοστάρ ας πούμε, στο Ανατολικό Μοστάρ, εκεί που ζουν ε, οι μουσουλμάνοι, μεταφέρθηκαν στο δυτικό τμήμα, χωρίς να τους εμποδίσει η αστυνομία. Κατέστρεψαν, πυρπόλησαν και η αστυνομία ε, τους κοιτούσε απλώς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, ακριβώς όπως είπαν και οι συνάδελφοι, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Και αύριο που θα έχουμε εδώ την κυρία Άστον, θα πρέπει να τη ζητήσουμε να μας πει πώς έχει η κατάσταση, ευελπιστώντας ότι θα καταλάβουμε κάτι περισσότερο και ότι θα καταστεί σαφές και στην Επιτροπή μας, αλλά και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, ε, το περί τίνος πρόκειται και ότι θα καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Βοσνία Ζεγοβίνη αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, ενδεχομένως να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα. Και εν τέλει να καταλάβουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις διαδηλώσεις. Γιατί δεν είναι μονάχα κοινωνικού περιεχομένου αυτές οι διαδηλώσεις. Οπωσδήποτε υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα που δικαιολογούν μια τέτοια κατάσταση, αλλά δεν είναι ε, ε, αυτή η ουσία του πράγματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε διάφορες γνωμοδοτήσεις σε σχέση με την απαλλαγή που αφορά την Κομισιόν για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε καταρχήν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια θετική γνωμοδότηση γιατί η υπηρεσία αυτή έχει εκτελέσει τον προπολογισμό της χωρίς το ελεκτικό συνέδριο να εντοπίσει ουσιώδη σφάλματα. Αυτό φαίνεται και στη γνωματοδότησή μου. Παρ' όλα αυτά <clears throat> κατατέθηκαν 14 τροπολογίες. Μερικές από τις δικές μου και άλλες. Βρήκαμε κάποιες συμβαστικές λύσεις η οποία καλύπτει πέντε από αυτές τις τροπολογίες. Θέλω όμως να τονίσω και πάλι και το λέω στη γνωμοδότηση ότι η επιλογή του, πληθυσ... του προσωπικού στα υψηλά κλιμάκια του, ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης είχε δεσανάλογα μικρό ε, αριθμό γυναικών. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό και γι' αυτό έχουμε δεχτεί τις τροπολογίες της κυρίας Γιατεμάχη, του κυρίου Μπίλαν και της κυρίας Βαϊντέρ. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι για τα κράτη-μέλη το να μπορούν να υπάρχουν αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένες χώρες όπου δεν υπάρχουν διμερείς αντιπροσωπείες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον τις πιο μικρές και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε την ε, υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια ευκαιρία και σαν ένα τρόπο εξοικονόμηση χρημάτων σε αυτού του δύσκολου ε, καιρού. Υπάρχει και η τροπολογία του κ. Σαλαφράγκα που ζητά να υπάρξει μια αντιπροσωπεία στον Παναμά που είναι μια χώρα κομβική για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λατινική Αμερική λόγω της γεωγραφικής θέσης του Παναμά στην ε, Κεντρική Αμερική μεταξύ των δύο τμήματων της ε, Αμερικανικής Υπήρου και έχουμε τονίσει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί και η ασφάλεια του προσωπικού της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης στο εξωτερικό όπως και η ασφάλεια των ε, επικοινωνιών τους. Νομίζω εν γέννη ότι οι δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από τη λειτουργία της Επιτρόπης Εξωτερικών Δράσεων για να υπάρχει μεγαλύτερη ακτινοβολία της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικές και γι' αυτό είναι απαραίτητο το στίχημα αυτό της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να ενισχυθεί με την καλύτερη κοινή δράση και το συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την υπηρεσία. Υπήρξε και εδώ μια συμβιβαστική τροπολογία που νομίζω ότι θα γίνει δεκτή από όλες τις πολιτικές απόψεις σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Μουνή πρώτα απ' όλα για τις δύο γνωμοδοτήσεις της που νομίζω ότι εγγράφονται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση και είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις κατευθύνσεις, με τις γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγή το να υπάρξουν σωστέ πολιτικέ και κυρίω η διαφάνεια στην χρήση και τη διαχείριση των πόρων του προπολογισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε να υπογραμμίσω τι σημασίε, τι δυσκολίε που αναφέρονται και στι δύο γνωμοδοτήσει για τι δραστηριότητε αυτέ που χρηματοδοτούνται μέσω άλλων διεθνών οργανισμών. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει σημαντικά ποσά σε άλλους διαχειριστές όπως είναι τα Έθνη και επομένως θα πρέπει και εκεί να πριτανεύουν οι αρχές της αποτελεσματικότητας και της προσθέμενης αξίας που είναι πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση αυτή αυτή, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μουνιέθ για το πνεύμα συνεργασία που έχει δείξει και η ομάδα μα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τι συμβαστικέ τροπολογίε που έχουν τύχει διαπραγμάτευση μεταξύ των καταθετών τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Μίλησα μονάχα για την πρώτη γνωμοδότηση για την ε, εξωτερική υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά έχουμε και την ε, απαλλαγή τη Κομισιόν. Έχω πάρει 10 τροπολογίε και έχω καταθέσει τρει τροπολογίε και εγώ και μια προφορική. Δεν νομίζω ότι αυτή η έκθεση δημιουργεί προβλήματα πέραν το γεγονό ότι υπάρχει από τι διάφορε ομάδε μια ε, κριτική εστίαση ισχυρότερη ή ασθενέστερη σε σχέση με τα σφάλματα τα οποία εντοπίστηκαν στο, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αυτά τα λάθη που αναφέρει το, το ελεγκτικό συνέδριο έχουν να κάνουν περισσότερο με τη μεθοδολογία δειγματοληψίας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια καλύτερη ε, μεθοδολογία σε σχέση με την ε, εκαθάριση των προκαταβολών. Επίσης υπάρχει και μια παράγραφος όπου ζητάμε να υπάρξει καλύτερη επαναχρησιμοποίηση του υλικού που χρησιμοποιείται στις ε, αποστολές εκλογικής παρακολούθησης που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και σε περαιτέρω αποστολές που ε, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μειώσουμε τα χρήματα τα οποία δίνουμε στις εκλογικές αποστολές ε, παρακολούθησης. Δεν χρειάζεται λοιπόν όλο το γραφειακό υλικό, όλο το πληροφορικό υλικό να αφήνεται στις χώρες αυτές, ένα τμήμα αυτού θα μπορούσε να δοθεί σε ΜΚΟ ή σε άλλους φορείς. Είναι όμως πολλές φορές δεκάδες υπολογιστών, εκτυπωτών που μένουν στη χώρα που έγινε η εκστρατεία που μενουν στη χωρα που ειναι η εκστρατεια παρακολουθησης και στην επόμενη διαδικασία εκλογική παρακολούθηση πρέπει να ξαναγοράσουμε αυτό το υλικό. Αυτό είναι μια δαπάνη την οποία μπορούμε να αποφύγουμε. επίσης υπάρχει μια μόνιμη έλλειψη επαρκούς προϋπολογισμού για τις ενέργειες της ε, παρακολούθησης αυτής και ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και οικονομικοί με τις δαπάνες μας ώστε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και σε μελλοντικού προϋπολογισμούς να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη επαρκών πόρων και πόρων επιμελητίας κυρίως στην Κομισιόν αλλά ιδίως και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μούνιες. Κυρία Γιάτεν Μάκη. Και μάλλον να σας πω κιόλας ε, καλό απόγευμα σε όλους σας, να σας χαιρετήσω μια και τώρα πήρα τη θέση του Προέδρου. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μουνίσε, με την οποία η ε, συνεργασία υπήρξε εξαιρετική. Ε, έχουμε κάποιες παρατηρήσεις βέβαια να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να γίνεται με ανοιχτό και διάφανο τρόπο η διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια βασική θεμελιώδης αρχή. Και νομίζω ότι εδώ δεν υπογραμμίζεται επαρκώς. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Ανησυχεί η ομάδα μου διότι οι διαχειριστές δεν ε, φαίνεται να γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες. Αυτό συνδέεται βέβαια με το προηγούμενο, ε, τη διαφάνεια και το άνοιγμα. Θα πρέπει να επαναστοχεύσει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι γνωστή να είναι γνωστοί οι όροι και να είναι γνωστό το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα από τους διαχειριστές. Τρίτον, ο αριθμός των ε, ε, υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, ε, μακράν υψηλότερος από τις υπόλοιπες υπηρεσίες και εδώ θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση. Επίσης, η γεωγραφική ισορροπία, δηλαδή όταν η εκπρόσωπος άρχισε την εργασία της μας είπαν ότι ε, θα διεσφάλιζε την καλή γεωγραφική ισορροπία. Δεν το είδαμε όμως και όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών και όσον αφορά την γεωγραφική ισορροπία δεν είναι καλά τα αποτελέσματα και εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά γιατί ε, δεν καταλαβαίνω πώς φτάσαμε εδώ τη στιγμή που δημιουργείται μία νέα διοίκηση, εξ ολοκλήρου νέα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν σε διοικήσεις ε, οι οποίες υφίστανται ήδη Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Ευχαριστώ. Προέδρο, ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κανεί το λόγο. Αν όχι, η κυρία Μουνή, αν θέλει να κάνει κάποιε τελικέ παρατηρήσει. Και εγώ φυσικά <clears throat> συμμεράζομαι την ε, ανησυχία για το μεγάλο αριθμό υψηλών στελεχών στην υπηρεσία εξωτερική δράση και την έλλειψη ε, ισορροπίας ε, σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο ισορροπία μεταξύ των φύλων. Τονίζω ότι η ισορροπία μεταξύ των φύλων πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη και αυτό αναφέρεται σαν ένα από τα βασικά σημεία ανησυχίας από τα μέλη της Επιτροπής μας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ίδιο ισχύει για την έλλειψη διαφάνειας. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερη έλεγχη και για την Κομισιόν και για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επομένως, συμμεριζόμαστε και τις επικρίσεις και υποστηρίζω και αυτές τις προτάσεις που θεωρώ ότι είναι πράγματι επικοδομητικές και πρέπει να ε, θεωρηθούν ότι είναι επικοδομητικές και δεν έχουν σαν στόχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μεγαλύτερη δυσπιστία των πολιτών στις πολιτικές εξωτερικής εξωτερικής και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να προχωρήσουμε σε πιο επικοδομητικά μέτρα και αυτό ακριβώς κάνω και εγώ με το να δεχτώ τις περισσότερες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τη συζήτηση για αυτά τα δύο θέματα. Να υπενθυμίσω τώρα στα μέλη ότι η ψηφοφορία για τα δύο θέματα θα γίνει αύριο το πρωί. Περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η χρήση της, ε, των ε, οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλείο της διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια σύσταση προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Δεύτερη εξέταση του σχεδίου σύστασης για την χρήση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ως εργαλείο διπλωματίας και προβλέπεται αύριο πρέπει να, γίνει ψηφοφορία και θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή τον Sir Graham Watson για να παρουσιάσει τη θέση του για τις τροπολογίες και τις ενδεχόμενες συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδελφούς και κυρίως τους και οδησηγητές για τη βοήθεια που μου παρέσχουν για αυτή την έκθεση. Και αύριο το πρωί θα ε, καταθέσουμε την έκθεσή μας προς ψηφοφορία στην Επιτροπή. Το κείμενο έχει εγκριθεί, το αρχικό κείμενο, και είμαι ευγνώμων στους σκιώδησηγητές για τον πολύ επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το θέμα. Νομίζω λοιπόν, Πρόεδρε, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ότι χρειαζόμαστε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν τις αξίες που έχουν κατοχυρωθεί στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα χρειαζόμαστε τα μέσα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις σχέσεις με τρίτες χώρες. Έχει, υπάρχει διαδεδομένο το συνέστημα ότι τα μέσα ενημέρωση σε διεθνές επίπεδο παίζουν αλλά και θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας τύπου, της ελευθερίας γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό που αναμένει κανείς από ευρωπαϊκή σκοπιά είναι ότι θα προσφέρουν αξιόπιστη εργασία, ε, θα σέβονται την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα της ε, δημοσιογραφίας. Γι' αυτό καλούμε το Συμβούλιο, την Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης και το Κοινοβούλιο να ορίσουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και αυτό ως τμήμα της στρατηγικής τους στις εξωτερικές τους δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δηλαδή. Ελπίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα επηρεάσουμε ένα θετικό κλίμα στις τρίτες χώρες για να αναπτυχθούν τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης και θα στηρίξουμε γενικότερα τα μέσα ενημέρωση σε ολόκληρο τον κόσμο έτσι ώστε όλα να προσχωρήσουν σε έναν παγκόσμιο χάρτη έτσι ώστε να ε, διασφαλίζεται η ουδετερότητα ανεξάρτητα από οποιοδήποτε ε, κυβερνητικό κόμμα, επιχειρηματίες, επιχειρηματικά συμφέροντα να ε, χρησιμοποιείται η τελευταία τεχνολογία για να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στα, ε, στην κοινή γνώμη. Και για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε να υπάρχει και ένας ε, χάρτης ε, των μέσων ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διευκρινίζει τις αξίες μας και θα προάγει την αντικειμενικότητα της ενημέρωσης. Χάρη της, ε, των παρεμβάσεων των συναδέλφων την προηγούμενη φορά είχαμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση σχετικά με την έδρα του Euronews και έχω κάνει τώρα μία πρόταση στην τροπολογία υπαριθμών 92 που λέει να ενισχυθεί η δυνατότητα, η αποτελεσματικότητα των Euronews στις Βρυξέλλες. Δεν πρέπει απαραίτητα να μεταφερθεί η έδρα τους στις Βρυξέλλες. Ε, οι δημοσιογράφοι μπορούν και πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο λήψη αποφάσεων για να έχουν ταχύτερη ενημέρωση και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη των υπολείπων κρατών σχετικά με το θέμα αυτό και αυτό πριν από την αυριανή ψηφοφορία. Μπορέσαμε να ε, ομαδοποιήσουμε σχεδόν όλες τις ε, άλλες ε, τροπολογίες. Έχουμε τώρα περίπου έξι συμβαστικές τροπολογίες και ελπίζω ότι τα μέλη θα στηρίξουν αύριο τις ε, τροπολογίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας έτσι ώστε το όλο θέμα να ψηφιστεί στην δεύτερη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κ. Πρέντα είναι ο σχεδιασμό τη της ομάδας μου, ο οποίος είχε μια δυσκολία για να μπορέσει να έρθει στις Βρυξέλλε. Θα έρθει αργότερα. Μου ζήτησε ενδιαμέσως να εκφράσω την θέση του εξ ονόματος του, της πολιτικής μου ομάδας προς τον κύριο Βότσον και τους άλλους και θέλω να εκφράσει, να εκφράσει την ικανοποίησή του για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαν στη συνάντηση των Σκιωδών στο Στρασβούργο. Η πολιτική μου ομάδα θέλει να εκφράσει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι υπήρξε μια σαφή σύγκληση απόψεων σε ό,τι αφορά στις πρωτοβουλίες που προτείνονται στο έγγραφο αυτοεργασίας και η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή την πρόταση σύσταση στο σύνολό του και επίσης να υποστηρίξει και τις εξτροπολογίες συμβασμού που έτυχαν διαπραγμάτευσης. Ο κύριος Πρέντα λοιπόν και εγώ ίδιος θεωρούμε ότι βελτιώνει σημαντικά το αρχικό κείμενο οι έξι αυτές τροπολογίες ε, συμβιβασμού και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη πλήρως οι προτάσεις και οι ανησυχίες της ομάδας μας μέσα από διάφορες τροπολογίες. Ο κύριος Πρέδα θέλει να εκδηλώσει ιδιαίτερα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΣΥΤΗΣ έχει διαφοροποίησει ελαφρώς την πρότασή του σε σχέση με την έδρα του Euronews, ξέροντας ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τη δική μας πολιτική ομάδα και επομένως οι τροπολογίες μας για το θέμα αυτό ελήφθησαν υπόψη. Τέλος, <clears throat> θέλω να εκφράσω την θέλει να εκφράσει την ικανοποίησή του ότι οι τροπολογίες μας 7, 8 και 11 ελήφθησαν υπόψη πάρα πολύ σοβαρά, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εξωτερικής υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικού χαρακτήρα για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα θέματα διαλόγου με τρίτες χώρες στα ζητήματα αυτά. Αυτές είναι λοιπόν η, τα σχόλια του κυρίου Πρέντα και θέλω να διαβιβάσω τον εισηγητή την θετική μας αντιμετώπιση σε σχέση με την έκθεση και την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θα να λάβει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντένις Μάρκερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μίλησαν, με πρώτον και καλύτερο βέβαια τον εισηγητή. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα, είδαμε και ενδιαφέρουσες τροπολογίες. Πιστεύω ότι οι πολιτικές ομάδες θα συμφωνήσουν ε, στο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, μια ενωσιακή στρατηγική δηλαδή. Ε, έχουμε μέσα ενημέρωσης τα οποία φυσικά θα πρέπει να διατηρήσουν την, την ανεξαρτησία τους, τη δυνατότητα αντίδρασή τους, την δυνατότητα επίσης να παρέχουν αντικειμενική και υψηλού επίπεδου ε, δημοσιογραφική πληροφόρηση. Στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε τον, ε, την αιτιολόγηση των ε, πράξεών μας, ε, προωθώντας ταυτοχρόνως τις αρχές και τα ιδεώδη της δημοκρατίας. Υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες. και είδαμε και τις υπόλοιπες τροπολογίες, μερικές είναι πιο αμφιλεγόμενες από άλλες όσον αφορά το τελευταίο στοιχείο, της αξίες ε, της ε, δημοκρατίας. Επ' αυτού υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το κείμενο πιστεύω ότι θα πρέπει να προσφέρουμε στη ε, στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινή γνώμη μία ενιαία ε, ε, ιδέα που θα βασίζεται στην, προς, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μην λησμονούμε ότι θα πρέπει να αποτελούμε παράδειγμα η ε, πολιτική μας, η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ε, αυτές ε, τις αρχές και μάλιστα να βασίζεται στις αρχές αυτές γιατί διαφορετικά θα χάσουμε την αξιοπιστία μας. Οι τροπολογίες μας δεν έγιναν εν συνόλο δεκτές και γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να ξανασκεφτείτε λίγο τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει στα πλαίσια της αυριανής ψηφοφορίας πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ε, μπορούμε να επιτύχουμε καλό αποτέλεσμα. Ο κύριος Τάνοκ δεν είναι εδώ, είναι ο σκιώδης για τους ε, συντηρητικούς, δεν είναι εδώ. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Βερζιά της Γκουε. Δεν βλέπω να είναι παρούσα. Επομένως επανέρχομαι στον εισηγητή. Σερ Γκράχαμ, θέλετε να πείτε δύο λόγια για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς ε, τον κύριο Σαλαφράκα, ε, Σαλαφράγκα καθώς επίσης και τους, ε, τον κύριο Ντένις Μάκερ για, τα όσα είπαν και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στην αυριανή ψηφοφορία έτσι ώστε να περάσει το θέμα να φτάσει στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση και από αυτού του σημείου. Όσον αφορά το αρχικό σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως, πρέπει να σας πω ότι η ψηφοφορία επί της εκθέσεως για την ολιστική προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβει χώρα την 17η ε, Φεβρουαρίου. Δεύτερο είναι ότι την ε, Τετάρτη θα γίνει συζήτηση στη ΣΕΔΕ. Τώρα, σύσταση προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την Εξωτερική Υπηρεσία, την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, όσον αφορά την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ιράν. Η κυρία Μουνής είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Θα θυμάστε ότι την 21η Ιανουαρίου οργανώσαμε και ακρόαση για το θέμα αυτό. Τώρα υπάρχει μια ενδιάμεση, έχει ολοκληρωθεί μάλλον ε, η ενδιάμεση συμφωνία ε, για την ε, πυρηνική ενέργεια τώρα λέω που αυτή η συμφωνία ε, έλαβε χώρα, χάρη κυρίως στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ο καταλληλότερος χρόνος για να ξεκινήσουμε συζητήσεις με το Ιράν. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει τα μάλα στην ε, κατάσταση αυτή μέσω της εξωτερικής της πολιτικής. Έχοντας πει αυτά, θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μουνής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην περίπτωση του Ιράν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ορόσημο της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής διπλωματίας και συγκεκριμένα της κυρίας Άστον, η οποία ενεπλάκει πάρα πολύ ενεργά στις προσπάθειες για να βελτιωθεί το σύνολο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν και <clears throat> τονίζω ότι αυτές είναι οι σχέσεις οι οποίες πρέπει να συνάδουν με την ε, το μέγεθος και την ισχύ του Ιράν και την θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει μια ισορροπία σε μια περιοχή που υπάρχουν πολλές αντίπαλες τάσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας μεγάλης, το επαναλαμβάνω και πάλι, διπλωματικής επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Τίποτα ακόμα δεν έχει εδρεωθεί, δεν υπάρχει καμία εγγύηση να συνεχίσουν τα πράγματα αυτά, αλλά βρισκόμαστε σε μια εκκίνηση μια κατάσταση η οποία είναι πολύ θετική και επομένω θα πρέπει να την υπογραμμίσουμε ότι είναι πραγματική θετική όπω αναφέρεται και στο σχέδιο αυτό έκθεση. Και έχει ανοίξει και η προθεσμία για τι τροπολογίε από του συναδέλφου που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτήν την ε, αξιολόγηση. Για τη σύσταση αυτή δεν πρόκειται μονάχα λοιπόν για κάτι το οποίο έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν οι εκλογέ του 2013 του Ιουνίου στο Ιράν, από τις οποίες προέκυψε μια σαφής αλλαγή προς το καλύτερο στο εσωτερικό του Ιράν, μια θετική εξέλιξη και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει και από αυτή την εσωτερική αλλαγή στο Ιράν να βελτιωθεί, να προκύψει μια βελτίωση για το ρόλο του Ιράν στη διεθνή κοινότητα. Η σύσταση αναφέρει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία καθώς και την θετική ε, στάση των ΗΠΑ και τη θέλησή τους, τη βούλησή τους για να βελτιωθούν οι σχέσεις τους με το Ιράν <clears throat> και να υπάρξει μια διαφορετική στάση σε σχέση με τις κυρώσεις. Αν οι κυρώσεις είχαν θετικό αποτέλεσμα ως τώρα, από εδώ και πέρα κινδυνεύουν να γίνουν αντιπαραγωγικές και να υπονομεύσουν την αξία της συμφωνίας της 20 Ιανουαρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα διαφορετικό σκηνικό πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του, να μην μείνουμε έξω από τη διαδικασία αυτή, η οποία είναι μια διαδικασία <clears throat> που έχει τονίσει την αξία της ευρωπαϊκής ε, διπλωματίας. Βασίζεται η σύστασή μας σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τα ποινικά θέματα, τον διάλογο για τα ποινικά θέματα πρέπει να αναπτυχθεί με το Ιράν. Φυσικά χαιρετίζουμε την Συμφωνία της Γενέβης, θεωρούμε ότι δεν, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα εναλλακτική από μια διαπραγματευμένη και ειρηνική λύση για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πλήρως οι ανησυχίες της ε, διεθνούς κοινότητας σε σχέση με τις δράσεις του Ιράν στα πληνικά θέματα και τον εμπλουτισμό ουρανίου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη στάση του Συμβουλίου και της ε, ΥΠΑ εκπροσώπου καθώς και των κρατών των ε, τριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τριών και των άλλων τριών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ όμως ο διάλογος αυτός πρέπει να έχει δύο πτυχές. Μία, αν θέλετε, μία οδό που βασίζεται σε δύο παράλληλα μονοπάτια. Ένα από τα βασικά θέματα που μα ενδιαφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ιράν είναι το θέμα τη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά το γεγονό ότι υπήρξαν βελτιώσει τον τελευταίο καιρό και υπήρξαν βελτιώσεις με τα πολιτικά δικαιώματα και η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά προβλήματα ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, θανατική ποινή, σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικέ και όχι μόνο μειονότητες, τις ομάδες των, ε, των ΛΟΑΔ, την επιβολή σε ανηλίκους της θανατικής ποινής, όλος αυτός λοιπόν ο διάλογος δεν πρέπει να ανασταλεί, ούτε πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας απλώς και μόνο επειδή επετεύχθη μια συμφωνία σε σχέση με τα ποινικά θέματα με το Ιράν. Το άλλο θέμα που ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο και αυτό είναι μια ιστορική διεκδίκηση πέραν των πυρηνικών θεμάτων είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε να επιμείνουμε για αυτό το θέμα. Και τρίτον, θελήσαμε να, να περιλάβουμε σε αυτή την ε, σύσταση να είναι σύντομη και συνοπτική. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε παραγράφους, να αναφερθούμε σε άλλα ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, αλλά εδώ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε μια γενική ανατομή του ρόλου του Ιράν στο παγκόσμιο στερέωμα, τη σχέση του με το Ιράν, με τη Συρία, συγγνώμη, τις ε, συγκρούσεις με άλλες χώρες, την ανάγκη να έχει ένα σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα πράξουμε γιατί είναι περιορισμένος περιορισμένη η έκταση μιας σύστασης. Θελήσαμε όμως από αυτή τη σύσταση να δημιουργήσουμε ένα επικοδομητικό κλίμα, να δώσουμε επικοδομητικά στοιχεία. Τονίζοντας ότι έχουμε τώρα νέες προοπτικές να προχωρήσουμε και πέραν των θεμάτων που είναι ιδιαίτερα επίμαχα με το Ιράν και να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια κοινή πολιτική, μια κοινή δράση με το εμπόριο ναρκωτικών. Παραδείγματο χάρη ξέρουμε ότι 80% των ναρκωτικών που έρχονται στην Ευρώπη περνάνε από το Ιράν και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και έχουμε ενώπιον μα ένα παράθυρο ευκαιρία για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ιράν σε επίπεδο επικοδομητικό και που δεν βασίζονται πια σε αμοιβέ απειλέ, σε αντιπαραθέσεις ή σε επιβολή κυρώσεων. Πρέπει λοιπόν να παροτρύνουμε τη διαδικασία αυτή διαλόγου με το Ιράν και διαπραγματεύσεων και ακριβώς σε αυτό επιμένει και η σύστασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ που θέλει να μιλήσει εξ ονόματος του κυρίου Ζαλεύσκη που είναι ο σκιώδης εισηγητής. Από ό,τι φαίνεται όμως όχι. Ε, κατόπιν τούτου θα ήθελα να δώσω λόγο στην κυρία Κρόμπερκ που εκτός του ότι είναι σκιώδης εισηγήτρια για τους πράσινους είναι και πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, της Αποστολής Αντιπροσωπής με το Ιράν. Έχετε το λόγο. Εμείς ε, καλωσορίζουμε αυτήν την έκθεση, είναι επίκαιρη. Ήταν απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί στη δουλειά που γίνεται από τη Σύναψη της Γενέβης. Και αυτή λοιπόν η έκθεση είναι πολύ σημαντική και για την κυρίαστον και για την παγκόσμια πολιτική. Επίσης ε, αντικατοπτρίζει και την ε, τις ε, προσδοκίες του Ιρανικού λαού, τη θετική αλλαγή. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει ε, να δεχόμεθα αυτό, αλλά να μην υπερβάλλουμε. Κατά τα άλλα, είμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο και είναι πολύ σημαντικό να εκφραστούν στην έκθεση ότι όλα τα κόμματα και ότι συμφωνούν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν εσκυρώσεις και οι Ιρανοί ε, θα πρέπει να επιτρέψουν πρόσβαση ε, σε όλες τις ε, στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Έχει φτάσει ποια στιγμή να έχουμε στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας σε τομείς όπου διαφωνούμε. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το διάλογο για θέματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα δικαιώματα. Έχουμε ε, τον Επίτροπο στα Ηνωμένα Έθνη, τον οποίο έχουν προσκαλέσει οι Ιρανοί μέχρι τώρα δεν του είχαν επιτρέψει την πρόσβαση και όταν λοιπόν μιλήσαμε με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν είναι προφανές ότι επιθυμούν να έχουν συζήτηση με τον εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν αυτό πρέπει να το προτείνουμε και είναι πολύ καλό το ότι η έκθεση ε, προβάλλει και την έννοια των ε, συγκρίσεων ε, σε σημεία αναφοράς γιατί νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να έρθουν πιο κοντά οι δύο πλευρές. Είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιβάλλει προσχεδιασμένα μέτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούει και την άλλη πλευρά και κυρίως όσον αφορά τη θανατική ποινή όπου το 80% αυτών των αποφάσεων έχουν ε, άμεση σχέση με τα ναρκωτικά. Οι Ιρανοί λοιπόν θέλουν να το ξανασκεφτούν το όλο θέμα και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τη συνεργασία με το Ιράν. Όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, όπως λέει και ο εισηγητής, ε, δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτή την ε, ισορροπία δυνάμεων με τη Σαουδική Αραβία. Πάντως αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι το Ιράν πρέπει να δείξει ότι έχει μια νέα εξωτερική πολιτική που θα δοκιμαστεί στην πράξη. Αυτή η έκθεση είναι το πρώτο βήμα. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλουν και πρέπει στο μέλλον να ανοίξουμε γραφείο στο Ιράν με έναν ειδικό συντονιστή ο οποίος ε, θα μπορούσε να ε, δώσει κάποια κίνηση στην όλη κατάσταση. Όταν επισκεφτήκαμε το Ιράν, όλοι οι πρέσβεις μας είπαν ότι είναι πραγματικά απόλυτα απαραίτητο να υπάρξει μια δική μας αντιπροσωπεία στο Ιράν. Κυρία Σάκη, ευχαριστώ πολύ. και τον εισηγητή αλλά και τους ε, συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Νομίζω πως ε, πράγματι είναι πολύ καλή η χρονική συγκυρία για να δούμε με επικοδομητικό αλλά και ανεξάρτητο τρόπο την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν, ε, γιατί έτσι πρέπει να ορίζονται οι σχέσεις αυτές. Θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε περισσότερα, αλλά το θέμα είναι με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μονάχα το θέμα της πυρηνικής ε, συμφωνίας. Στην ε, επίσκεψη που κάναμε το Δεκέμβρη ε, κατηδείχθη ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα και άλλων θεμάτων διεύρυνσης ας πούμε της αντιπροσώπευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης καταπολέμηση των ναρκωτικών, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πράγματα δηλαδή τα οποία οπωσδήποτε μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη ζωή των ε, στρατιωτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που βρίσκονται στο Αφγανιστάν. Επίσης, μεγάλος χώρος υπάρχει ακόμα και για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι αξίες καθολικές και παγκόσμιες που πρεσβεύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πω προς τα που θα κατευθυνθούν οι τροπολογίες μου. Πρώτον, ε, υπήρξε περιορισμένη δυνατότητα επιλογής ε, στις ε, εκλογές. Ε, επίσης ε, υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι έχουν ακόμα πιο επιθετική στάση απέναντι στις ε, ανοιχτές σχέσεις του Ιράν με τον, εξω, τον κόσμο σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε και τις συνεχείς και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν περίπου 1.700 εκτελέσεις κάθε χρόνο σε αυτή την Ισλαμική Δημοκρατία όσον αφορά το ζήτημα της συνεργασίας επί σειράς θεμάτων, πιστεύω πως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και την ε, συνεργασία καθώς επίσης και την ε, σταθεροποιητική δράση ε, που μπορεί να έχει η συνεργασία με τους Χεσμπολά Μπορούμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών καθώς επίσης ε, και τον ιδιωτικό τομέα και πιστεύω ότι οποιαδήποτε συνεργασία προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, εμπορίας ε, ναρκωτικών οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ε, δυνατότητα ε, δίκαιης δίκης ε, των υπόπτων καθώς επίσης και την κατάργηση της θανατικής ποινής για εγκλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε, να αναφέρουμε και αυτήν την διακυβερνοβουλευτική χάρτα την οποία υιοθέτησε το, ε, προσπέγραψε μάλλον το Ιράν το 1996 να αναφερθούμε εις τα δικαιώματα των μειονοτήτων, κυρίως της μειονότητας των ΣΥΧ, την δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο και με δικηγορική ε, αρρωγή, γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις όπου όχι μόνο δεν υπάρχει πρόσβαση σε δικηγόρο ε, και σε δίκαιη δίκη, αλλά εκδίδονται καταδικαστικές ή ακόμα και θανατικές ε, καταδίκες χωρίς να γνωρίζει καν η οικογένεια περί τίνος πρόκειται. Συμφωνώ ε, με τον προέστατο συνάδελφο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, ζητήσουμε και από την ύπατη εκπρόσωπο να ξεκινήσει συζητήσεις με την Ιρανική πλευρά. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία. Ε, τα οποία θα περιλαμβάνουν οι τροπολογίες μου. Οπωσδήποτε θα ήθελα να καλέσω όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ε, έκθεση γιατί πραγματικά πρόκειται για μια κατάσταση εξαιρετικά ευαίσθητη, είναι πολύ τρωτή και επομένως ε, πιστεύουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του έτσι ώστε να παραμείνουν οι δύο επικοινωνία ανοιχτοί με το Ιράν. Ο κύριος Μπέλτερ τώρα από την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ διάβασα το κείμενο αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα την ευκαιρία ήδη να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα και κατανοώ ποιες είναι οι δυσκολίες του έργου της Επιτροπής μας. Δεν θέλω να σας ε, κρύψω τις ανησυχίες μου σε σχέση με τα πυρηνικά θέματα στο Ιράν. Όταν μιλάτε για μεγάλες επιτυχίες, εγώ νομίζω πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να έχουμε επιφυλάξεις και ανησυχίες σε σχέση με αυτή τη συμφωνία και γενικότερα σε σχέση με την διεθνή πολιτική που ακολουθεί το Ιράν. Νομίζω ότι με τον πρόεδρο Ρουχάνη ορισμένα πράγματα έχουν <clears throat> επιδεινωθεί και έχουμε μεγάλες ε, ανησυχίες οι οποίες θα μου οδηγήσουν να καταθέσω κάποιες τροπολογίες. Μερικά σύντομα σχόλια. Μιλήσανε οι συνάδελφοι για το πρόβλημα της ε, διακίνησης ναρκωτικών που διέρχονται από το Ιράν και του προβλήματος της ε, τοξικομανίας στην Ιρανική κοινωνία και στην Ευρώπη το αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Η επαναστατική φρουρά στο Ιράν που είναι η σπονδυλική στήλη του καθεστώτος είναι έμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενοι στο εμπόριο ναρκωτικών. Επομένως είναι έμεσα η αμεσα εμπλεκόμενη στο εμποριο ναρκωτικων επομενως αιτία του προβλήματος. Υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις και με το Αφγανιστάν. Όταν μιλάμε για το Αφγανιστάν το Ιράν για πολύ καιρό είχε ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων από το Αφγανιστάν και υπήρξαν σε εφημερίδες πρόσφατα πολύ καλές αναλύσεις για το τι κάνει το Ιράν για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης από το Αφγανιστάν. Μιλάμε για ενδεχομένως και εκατομμύρια ατόμων. Αυτό το οποίο είδα στις ειδήσει αυτές είναι ότι το θέμα των ε, προσφύγων από το Αφγανιστάν είναι ένα είδος γεωπολιτικού παιχνιδιού που παίζεται μεταξύ της Τεχεράνης και του Καμπούλ. Έχουν χρησιμοποιηθεί σαν πιόνια σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι, κάτι το οποίο έχει πολύ αλληλεγγύες συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο για αυτούς τους πρόσφυγες. Αν δει κανεί λοιπόν πώ λειτουργεί η Ιρανική κοινωνία, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προβλήματα τα οποία θα μπορούσε κανεί να αναφέρει σε αυτή την έκθεση. και η αλλαγή του καθεστώτος δεν νομίζω θα αλλάξει πολλά πράγματα. Λένε πολλοί ότι είναι πιο διαπεφωτισμένος ο νέος πρόεδρος Ρουχανή σε σχέση με τους προκάτοχούς του, αλλά θα έχει να αντιμετωπίσει αντιπαλότητες από την, από την πολιτική τάξη. Δεν ξέρουμε λοιπόν αν θα μπορέσει να υπάρξει πρόοδος στην Ινδία, στην, στο Ιράν συγγνώμη, που θα βελτιώσουν και την κατάσταση εκεί. Ο πληθυσμός στο Ιράν κινδυνεύει να υποφέρει ακόμα και στο μέλλον. Ελπίζω ότι οι τροπολογίες που θα καταθέσουμε λοιπόν θα λάβουν υπόψη την πραγματική κατάσταση στη χώρα αυτή και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να πούμε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν το Ιράν σαν σε εταίρο, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το Ιράν είναι έτοιμο να παίξει το παιχνίδι μαζί τους και να τηρήσει τα κριτήρια τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Εγώ βλέπω αυτό το παιχνίδι σαν ένα επικίνδυνο παιχνίδι και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ακόμα μια αναλλακτική λύση, ενδεχομένως και τη χρήση στρατιωτικής βίας. Ευχαριστώ κύριε Μπέλτερ. Μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, εκτός και αν θέλει η συγγήτρια να πει κάτι. Παρακαλώ κύριε Μουνιές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε Μουνιέ. Ο κύριος Σαλαφράγκα ήθελε να πει κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο. Αλλά ο κύριος Σαλέσκι μου έδωσε μόλις ένα μήνυμα ως και ο της ομάδας μου που είπε ότι δεν θα μπορέσει να είναι παρόν εδώ λόγω κολλημάτων προεκλογικής εκστατείας στη χώρα του και απλώς ήθελε να τονίσει ότι θεωρεί ότι αυτό το σχέδιο σύστασης είναι μια καλή εκκίνηση, ένα καλό σημείο εκκίνησης Πιστεύω ότι και αυτός πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου <clears throat> έλαβαν χώρα 40 εκτελέσεις με απαγχωνισμό και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε είναι απαραίτητο να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση των διαφόρων πτυχών που υπάρχουν στη σχέση μας με το Ιράν. Πράγματι υπήρξε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις Τη Γενέβη για τα ποινικά θέματα, αλλά είναι μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα πρέπει να επιχειρωθεί στη συνέχεια και από αυτή την άποψη θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της εισηγήτριας στην ανάγκη, όπως μου λέει ο κ. Σαλεύσκη, να ενισχύσουμε το κεφάλαιο σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπε η κυρία Σάκε, ότι θα πρέπει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια ανεξάρτητη στάση για τα θέματα αυτά. Για μένα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εγγράφεται πλήρως στο πλαίσιο των ενεργειών, των επιτυχημένων ενεργειών που είχε η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει αποφασιστικά να υποστηρίξουμε τι επιτυχίε των κρατών μελών και τη Υπηρεσία Εξωτερικών Εξωτερική Δράση και φυσικά ως θεσμικό όργανο που υποστηρίζει ανέκλητα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά και με αυτό τρόπο την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και πρώτα απ' όλα να εξασφαλιστεί η προξενική θεώρηση για τον ειδικό εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να παραδοθεί από το Ιράν το ταχύτερο δυνατό. Αυτά είναι τα σχόλια του κ. Ζαλεύσκη σε σχέση με την ανάγκη να ενισχυθεί λιγάκι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύσταση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μουνίτη, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω σε όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο και έκαναν σχόλια για το κείμενο αυτό που είναι φυσικά ανοιχτό σε κατάθεση τροπολογιών. είναι ορισμένα πράγματα προφανή. Δεν έχουμε μια χώρα που πέρασε από τον άξονα του κακού στον παράδεισο των ε, χωρών που είναι κολοφόνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε μια διαδικασία, μια θετική διαδικασία, τουλάχιστον στην έναρξή της, αλλάζει η τάση που επικρατούσε μέχρι τότε, που είχε οδηγήσει το Ιράν να είναι εκτός της ε, ε, διεθνούς κοινότητος, λόγω και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά λόγω και του πυρηνικού, προβλ... πυρηνικού θέματος. Νομίζω ότι ο κύριος Μπέλτερ δεν μπορεί να αρνηθεί την πραγματικότητα ότι υπήρξε μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής ε, Διπλωματίας και των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να τονίσουμε φυσικά ότι είναι εύθραυστη αυτή η διαδικασία, όπως είπε και η κυρία Σάχη, και ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε κατά κάποιο τρόπο υποτιμητική ή συγκαταβατική με το Ιράν, απλώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια σειρά συντελεστών και στοιχείων που μπορεί να αλλάξουν τη θέση του Ιράν έναντι της διεθνούς κοινότητας. Οι κυρώσεις που ασκούνται κατά του Ιράν δεν είναι μονάχα το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικού των ε, ηγετών του Ιράν, αλλά υπάρχει και η απαγόρευση εισαγωγή πετρελαίου από το Ιράν που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν <clears throat> είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και για το πυρηνικό θέμα στην έκθεση αυτή υπογραμμίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόοδος και το ίδιο στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτά που λέει η κυρία Σάκε, Νομίζω ότι στην αιτιολογική σκέψη ε λέμε ότι εφόσον η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν χαρακτηρίζεται ακόμα από συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος να το πούμε πιο σαφώς. Υπάρχει μια συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και στη συνέχεια σε διάφορες παραγράφους της σύστασης αναφέρονται στο θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά το γεγονό ότι το έναυσμα για αυτή τη σύσταση ήταν η αλλαγή τη κατάσταση σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά, ένα μεγάλο μέρο τη σύσταση αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λυπηρό το γεγονό ότι υπήρξαν πολλέ εκτελέσει με τη νέα αυτή κυβέρνηση, με πρώτα τον κύριο Ρουχανή. Υπάρχουν πολλοί ε, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται ακόμα στη φυλακή. Αλλά οι θανατικές ποινές και οι εκτελέσεις έχουν να κάνουν με τη δικαστική εξουσία και όχι με τον πρόεδρο και είναι γεγονός ότι στη δικαστική εξουσία εξακολουθούν να υπάρχουν σκληροπυρηνικοί, συντηρητικοί, οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθμίσουν την αλλαγή πορείας για τα πυρηνικά θέματα, κρατώντας μια σκληρή γραμμή σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να καταδικάσουμε την πολιτική πορεία που έχει ξεκινήσει ο Ρουχανή η οποία είναι θετική γιατί αυτοί οι οποίοι είναι οι αντίπαλοι του Ρουχανί στο Ιράν θέλουν να κρατήσουν μια αντίθετη θέση με τη δικιά του στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απλώς πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Αλλά δεν πρέπει να περιορίσουμε τις δυνατότητες του Ιράν και να καταλογίζεται στο Ρουχανή ο οποίος είναι αυτός που ξεκίνησε τη διαδικασία αλλαγής στο Ιράν να του καταλογίζουμε τις ενέργειες αυτών που δεν υποστηρίζουν την αλλαγή. Και κύριε Μπέλτερ, είναι θέμα αξιοπιστίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην προηγούμενη έκθεση για το Ιράν εγώ ήμουν σκιώδης εισηγήτρια και εδώ έχουμε τους περιορισμούς χώρου και δεν μπορούμε να αναφέρουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα έχουμε εγκρίνει την προηγούμενη εβδομάδα μια έκθεση για τη Σαουδική Αραβία όπου έχει απαλληφθεί η παράγραφος που ζητούσε από τη Σαουδική Αραβία να βελτιώσει την νομοθεσία της και την πρακτική της σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά θέματα και απαλήφθηκε επίσης και η φράση που λέει ότι δεν υπήρχε θρησκευτική ελευθερία στην Σαουδική Αραβία. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές είναι χειρότερα τα πράγματα σε σχέση με το Ιράν. Όταν έχουμε δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μια περιοχή που είναι πυρίτιδα αποθήκη και υπάρχει μια περιφερειακή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χώρων αυτών που είναι οι δύο άξονες της περιοχής σε περιφερειακό επίπεδο στον αραβικό χώρο, δεν μιλάω τώρα για το Ισραήλ, στο μουσουλμανικό κόσμο γιατί το Ιράν δεν είναι αραβική χώρα. Και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε θετικά την Σαουδική Αραβία, ενώ στο Ιράν φαινόμαστε μαξιμαλιστές. Γιατί δεν αναφέρουμε, παραδείγματος χάρη, την ε, ε, <clears throat> καταπίεση της κοινότητας των Μπαχάη στο Ιράν. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν να είμαστε αντικειμενικοί, όχι ιδιαίτερα ήπιοι, όχι ε, εφεκτική με το Ιράν ή με τη Σαουδική Αραβία, αλλά πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια περιφερειακή αντιπαράθεση και πρέπει να κρατήσουμε μια ισορροπημένη θέση. Δεν είναι το Ιράν που είναι το κακό και άλλες χώρες που είναι καλές και το Ιράν έχει να αντιμετωπίσει λοιπόν τους συντηρητικούς, τους ε, σκληρούς δεξιούς. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν και εκεί μια σκληροπυρηνική στάση, ιδίω στη Γεωργία, η οποία έχει ξεπεραστεί. Θέλαν πολλοί να επιβάλλουν κυρώσεις και ουσιαστικά να σταματήσουν αυτή την ευάλωτη διαδικασία <clears throat> βελτίωση των σχέσεων με το Ιράν. Δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλου. Πρέπει παρόλα αυτά να είναι αρκετά απαιτητικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα πυρηνικά θέματα, αλλά να παροτρύνουμε τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις για τα ποινικά θέματα και παροτρύνοντας το Ιρανικό καθεστώς ή τουλάχιστον το τμήμα αυτού του καθεστώτος το οποίο έχει μια ακόμα αρνητική στάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αλλάξει την προσέγγιση του και να υποστηρίξει την αλλαγή στο Ιράν. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μουνίθ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτού του σημείου της μεριστείας διατάξεως. Προθεσμία για, την, ε, για τις τροπολογίες ε, είναι ε, η επόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Ο κύριος Χόβιτ είναι εδώ. Επομένω μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του επόμενου θέματο που αφορά τον περιφερειακό ρόλο του Πακιστάν και τι πολιτικέ του σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη έχουμε συζητήσει το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ζάλα τον Δεκέμβριο του 2013 και θα ήθελα να δώσω τον λόγο αμέσως στον κύριο Χόουιτ έτσι ώστε να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ζητά συγγνώμη από τον συνάδελφό μου που δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα και θα ήθελα να σας παρουσιάσω εγώ την εκθεσή του. Το κάνω αυτό με μεγάλη μου χαρά γιατί ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το Πακιστάν και έχω ε, συμμετάσχει πέρυσι στην σχετική αντιπροσωπεία την Γιουλάτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω και άλλους συναδέλφους βέβαια που συμμετείχαν και που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το Πακιστάν και με μεγάλη τους χαρά ε, συνεισέφεραν στην έκθεση του εισηγητή Ζάλα. Ε, το βασικό μήνυμα είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση. Ε, γίνεται αναφορά σε εκλογές του περασμένου έτους. Είναι η ήρεμη μεταφορά δύναμης για πρώτη φορά γίνει αυτό σε αυτή τη χώρα και αναφέρει στην έκθεσή του εισηγητή ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι διμερείς σχέσεις με αυτή τη χώρα. Ε, γνωρίζουμε ότι το Πακιστάν έχει στρατηγική σημασία. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρώπη να αρχίσει ε, τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν, την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και όπλων στο Πακιστάν υπάρχει ο κίνδυνος του εξτρεμισμού, γι' αυτό πρέπει να ε, διασφαλιστούν οι δημοκρατικές ε, διαδικασίες, ε, κυρίως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κοινωνικής αποστέρησης, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως φαντάζεστε, η έκθεση εκφράζει την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τους δημοκρατικούς θεσμούς, κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα και οτιδήποτε άλλο θεωρούμε σημαντικό. Στην έκθεση λοιπόν ο εισηγητής αλλά και όλοι μας ε, συστήνουμε τη βοήθεια στο Πακιστάν. Βεβαίως ε, Πρόσφατα αυτό επιβεβαιώθηκε στην Ολομέλεια και η έκθεση λέει ότι οι διμερείς σχέσεις θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ πιο πέρα από τις ανθρωπιστικές επαφές, να περάσουν στην ασφάλεια, στη συνεργασία και σε άλλα θέματα, έτσι ώστε να μπορούμε να προσβλέπουμε σε πιο πολιτικές σχέσεις με το Πακιστάν, να δίδεται προτεραιότητα συνεργασίας ε, με τη χώρα αυτή, ε, στη χώρα να υπάρχει βέβαια καλή διακυβέρνηση και να διδραματίζει χώρα επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή. Πρόεδρε, 58 είναι τροπολογίες για αυτήν την έκθεση. Εκ μέρους του κύριου Ζάλα θέλω να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς ε, με τις περισσότερες από αυτές τις ε, τροπολογίες. Στηρίζουμε τις ε, περισσότερες εξ αυτών. Υπάρχει ένας κατάλογος ψηφορίας και ο συγκητής πιστεύει ότι πολλές από τις τροπολογίες θα εμπλουτίσουν την έκθεση. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που υπάρχει ουσιαστική συνένεση ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες για αυτή την έκθεση. Έχω καταθέσει και εγώ εκ μέρου του πέντε συμβαστικέ προτάσεις που καλύπτουν κυρίως ευαίσθητα θέματα όπως την πυρηνική διάδοση, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν όμως εύκολο σχετικά να το συμφωνήσουμε αυτό οι σκιώδεις ηγητές. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι το επίμαχο όταν αυτά όλα θα ψηφιστούν στην Επιτροπή. Και θέλω να ολοκληρώσω ευχαριστώντας ε, τους και ηγητές για τη θαυμάσια συνεργασία με τον κύριο Ζάλα για τις ε, τροπολογίες τους. Νομίζω αύριο το πρωί ε, δεν θα υπάρξει καμία συζήτηση και βεβαίως μέχρι τότε περιμένω με χαρά τις ερωτήσεις σας και θα κάνω ό,τι μπορώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γκάλα, τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο κύριο Ζάλα για την έκθεση αυτή που είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Η έκθεση αυτή ρίχνει φως σε όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για τις εξελίξεις στο Πακιστάν αλλά και γενικότερα στην περιοχή όπου βρίσκεται αυτή η χώρα. Η έκθεση παρουσιάζει με σαφήνεια τις δυνατότητες συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πακιστάν. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε ένας σημαντικός εταίρος για το Πακιστάν ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά την άποψή μου ε, σωστά ε, προβάλλονται η συνεργασία σε αναπτυξιακά θέματα. Αυτό έτσι λέγεται γιατί κυρίως βεβαίως πρόκειται εδώ για θέματα παιδείας, παιδεία, παιδεία και πάλι παιδεία. Συνεργασία πρέπει να υπάρχει και στην προαγωγή της δημοκρατίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και εγώ μπόρεσα να συμβάλλω κατά τη σε αυτό το θέμα όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο με συμμετοχή σε ε, αποστολές παρακολούθησης ε, εκλογών, αλλά και το τι έγινε μετά τις εκλογές. Έχουμε το GSP από τις αρχές αυτού του έτους και έτσι λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθούν περαιτέρω οι εμπορικές σχέσεις. Υπάρχουν βέβαια και οι προϋποθέσεις ε, να υλοποιηθούν και όλα αυτά που έχουν σχέση με το GSP Plus ε, και έχουν σχέση με το εργατικό κυρίως δίκαιο, τη μη διακριτική μεταχείριση των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών. Κατά την άποψή μου λοιπόν όλα αναφέρονται μια χαρά Υπάρχουν βέβαια κάποιες δικές μας ε, μικρές ε, παρατηρήσεις, παραδείγματο χάρη ένα θέμα του ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στο Πακιστάν και την Κίνα. Και βέβαια πρέπει να σταθεροποιείται η περιοχή. Ε, και όταν έχουμε έτσι μια δευτερεύουσα πρόταση που να λέει should not undermine, δεν πρέπει να υπονομεύει δηλαδή, είναι σαν να ε, λέμε στους ε, Πακιστανούς ότι κοιτάξτε στις σχέσεις με τους Κινέζους έχετε τη δυνατότητα να υπονομεύσετε την κατάσταση σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα στον συνάδελφο κάπως να το υποβαθμίσει αυτό, απλά να κάνει λόγο για την βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή, κάπως έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Κατά τα άλλα, εμείς στηρίζουμε τους πέντε συμβασμούς που έχουν διατυπωθεί και κυρίως ε, τον συμβασμό υπαρθμών 2 στη νέα του διατύπωση. Αυτό είναι σημαντικό για μένα και θέλω να το υπογραμμίσω. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ Μιχαήλ. Και τώρα ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μιχάλα Ράιτ, εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Um, uh, Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω την άποψή μου. Καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή και κυρίως ε, την ε, ε, δυνατότητα, την ευκαιρία που δίνεται στο Πακιστάν να αναπτύξει περιφερειακό ρόλο. Όντως στην έκθεση αυτή αναφέρονται τα κυριότερα ζητήματα. Η αναφορά στην διακοινοβουλευτική διάσκεψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια καινοτομία η οποία δίνει την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει το ε, διάλογο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τις ε, συμφωνίες ε, και συνθήκες οι οποίες αφορούν την εργασία και τα λοιπά. Και επομένως να υπάρξει πραγματικά οικονομική μεγένθηση για το Πακιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επανειλημμένα έχει διατυπώσει, ενδιαφέρεται και δεσμεύεται απέναντι στο ε, Πακιστάν έτσι ώστε να αναδειχθεί ο ζωτικός ρόλος που παίζει το Πακιστάν στην ευρύτερη περιοχή. Κατά αυτή την έννοια φρονούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλες μάλλον θα πρέπει να δραχθούμε όλων των ευκαιριών ε, έτσι ώστε ε, να αναπτύξουμε τις σχέσεις με το Πακιστάν και έτσι ώστε ε, να υπάρξει πραγματικά ειρήνη αλλά και οικονομική ανάπτυξη στο Πακιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Richard, um, Κύριε Σιώη, πάρα πολύ σύντομος μπορώ να είμαι. Ε, βεβαίως είμαι ανοιχτό σε όλα τα σημεία του ε, κύριου ε, ε, Κάρλος. Όσον αφορά την τροπολογία 31 του, των Πρασίνων και την τροπολογία 32, ε, δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν μια προφορική τροπολογία αύριο, ναι, θα μπορούσα να την δεχτώ. Και θα σκεφτώ όλα αυτά τα σημεία τα οποία έθιξε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, πάρα πολύ ωραία. Η επόμενη ανακοίνωση είναι ότι αύριο το πρωί θα λάβει η χώρα η ψηφοφορία επί της εκθέσεως αυτής. Μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε την ε, ε, μελέτη αυτού του σημείου και να πάμε στο επόμενο, το οποίο αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κόσμο πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών. Είναι μια έκθεση της συναδέλφου μας κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου. Και θα της δώσω αμέσως το λόγο. Μαριέτα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η έκθεση αυτή βέβαια ε, έχει προσλαμβάνει εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης κατά τις τελευταίες δεκαετίες ε, όπου έχουν αναδειχθεί θρησκευτικές και πολιτιστικές διαφορές σε πολιτικούς παράγοντες. Ε, οι αξίες και οι αρχές της Ένωσης βέβαια πάντοτε υπήρξαν ανεξίθρησκες και ανεξάρτητες από τις πολιτιστικές διαφορές και κυρίως πάντοτε έτειναν ε, στο να απομακρύνουν τέτοια ζητήματα από την άσκηση της πολιτικής. Δηλαδή πάντοτε υπήρχε μια αντικειμενικότητα η οποία βασίζεται κυρίως ε, στις αρχές και στις αξίες της Ένωσης που θέλουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξάρτητα από φύλλο, φιλή, θρησκεία, εθνική προέλευση κτλ. να ισχύουν το ίδιο για όλους. Ε, η έκθεση σας θυμίζω ότι τονίζει ποιες είναι οι αρχές επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή πολιτική της Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος της Ένωσης βέβαια στα πολυεθνικά φόρα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που προέρχονται από τις θρησκευτικές ε, διαφορές και τις επιρροές ε, στο διεθνές, ε, στη διεθνή πολιτική αρένα και βέβαια ποια είναι η αξιοπιστία και η συνεκτικότητα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Υπήρξε μία σειρά τροπολογιών από τους συναδέλφους και εργαστήκαμε μαζί και έχουμε παρουσιάσει 15 τροπολογίες συνδέοντας τις διάφορες τροπολογίες συναδέλφων Βεβαίως παρέμειναν και τροπολογίες οι οποίες δεν μπήκαν στις ε, συμβιβαστικές. Είχαμε μείνει από τη συζήτηση με τους ε, ε, σκιώδεις εισηγητές στο να τους αποστείλω μία τροπολογία ακόμα που αφορούσε την παρουσία και την κατάσταση των χριστιανών στις τρίτες χώρες ε, για την οποία υπήρχαν αρκετές τροπολογίες και έπρεπε να γίνει συνδυασμός. Εγώ απέστειλα και αυτή την τροπολογία 16 ε, στους συναδέλφους, η οποία έχει ως εξής ε, εκφράζει την ανησυχία, μάλλον θα σας το πω στα αγγλικά, expresses its concern over proliferation. Εκφράζει την, ανησυχία, εκφράζει την ανησυχία της για την εξάπλωση της μυσαλλοδοξίας και ζητά πολλέ θρησκευτικέ κοινότητε μεταξύ των οποίων τον, τους χριστιανούς να εξασφαλίσουν την ε, θρησκευτική ελευθερία και ιδίως χριστιανούς που οι οποίοι σε πολλές χώρες λόγω της πίστης τους υφίστανται κατά πίεση και επίσης καταδικάζει τις προσπάθειες να κλείσουν εκκλησίες στον κόσμο. Ε, ε, δεν συμφωνεί με την τροπολογία αυτή ε, ενώ η ε, σοσιαλιστική ομάδα συμφωνεί καθώς και η Έκρες συμφωνεί. Αυτές είναι οι 16 τροπολογίες. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι ε, οι χριστιανοί αναφέρονται απλώς και ελάχιστα, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην κατάσταση που υπάρχει στις διάφορες χώρες και να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν θεωρούμε ότι μόνο οι χριστιανοί έχουν υποστεί διώξεις βέβαια σε διάφορες χώρες αλλά κυρίως σε αυτή τη φάση και στην Αφρική και χωρίς να αναφέρουμε χώρες και στην ε, Μέση Ανατολή ε, έχει υπάρξει ε, μία εντονότατη καταδίωξη των χριστιανών και η αναφορά αυτή το Including Christians είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στην έκθεση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια λεπτή υπόθεση, χωρίς αμφιβολία, αλλά πιστεύω ότι η έκθεση έχει δομηθεί έτσι, αλλά και οι τροπολογίες των συναδέλφων, ώστε να μην θεωρηθεί ότι είναι μια έκθεση μεροληπτική, η οποία κατά κάποιο τρόπο θέλει να υποστηρίξει ότι η μόνη θρησκεία πρέπει να την χάνει σεβασμού είναι ο χριστιανισμός κλπ. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει μέσα στην έκθεση. Υπάρχει αρκετή αντικειμενικότητα και νομίζουμε ότι μπορεί να ειδωθεί με την αντίστοιχη ε, αντικειμενικότητα και από τους τρίτους παρατηρητές και από τις άλλες χώρες. Βεβαίως, αυτό που στην ουσία διαφαίνεται από την έκθεση είναι ότι οι πολιτιστικές και θρησκευτικέ διαφορές δεν μπορούν να γίνουν δικαιολογία για βιαιότητες και παραβιάζεις των ατομικών δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο που αυτό ισχύει και στην δική μας ευρύτερη περιοχή, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των συναδέλφων επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ Μαριέτα. Θα δώσω το λόγο στην κύριε Λούτσεβα από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι ο πολιτισμός και τα θρησκευτικά θέματα είναι τελείως διαχωρισμένοι χώροι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και δεν έχουν καμία σχέση με την εξωτερική πολιτική. Η έκθεση αυτή καταδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Κατά την απόψή μου είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση, ιδίως μέσα στο πλαίσιο της τωρινή κατάστασης που έχουμε σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ένα παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο <clears throat> και γι' αυτό το λόγο η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ως προς το περιεχόμενό της, γιατί αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα, είναι έναυσμα για πολιτική προβληματική σε σχέση με τα θέματα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να εξετάσουν πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με τον καλύτερο τρόπο ένα κλίμα που να εξασφαλίζει τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε βέβαια διαφορετικές πολιτικές θέσεις, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία με την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές ήταν πάρα πολύ θετική και επίσης συζητήσαμε το θέμα αυτό στις πολιτικές μας ομάδες και υπάρχει μια ευρεία υποστήριξη από τη δική μας πλευρά των ε, τροπολογιών, των συμβαστικών ιδίω τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να καταδείξουμε την προσήλωσή μας για τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών και επομένως μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η αναγνώριση της θρησκευτική και εθνοτικής διαφορετικότητος. Έχουμε πάρει τις τελευταίες τροπολογίες, κάπως καθυστερημένα, αλλά έχουμε καταφέρει να τις ε, εξετάσουμε. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια ε, όξυνση των ε, διαφορών που υπάρχουν μεταξύ εθνοτικών ομάδων και θρησκευτικών ομάδων και ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πίεση κατά των χριστιανικών, κατά των χριστιανών. Με τις τροπολογίες αυτές είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται κατά οποιασδήποτε μορφής ακεροφροσύνης και εξτρεμισμού και κατά ομάδων οι οποίες δρούν με τρομοκρατικό τρόπο και φυσικά δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψει να αγωνίζεται για ένα πολύ δύσκολο μεν στόχο, αλλά σημαντικό να υπάρξει μια ενιαία κατάσταση σε σχέση με τις θρησκείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι την τελική ψηφοφορία και η ομάδα μας θα επανεπεξεργαστεί την έκθεση αυτή, αλλά εν γέννη και σε μεγάλο βαθμό υποστηρίζουμε την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία είναι αύριο. Ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η τροπολογία αυτή που μας διάβασε είναι καλό να συμπεριληφθεί. Κοιτάξτε, η έκθεση αυτή θέλει να αποσαφηνίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία ε, προώθηση οποιασδήποτε μορφής ε, ριζοσπαστισμού ή φανταμενταλισμού. Όσον αφορά τον συμβιβασμό 13, εκεί που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει ε, την ε, ανοιχτή ερμηνεία των θρησκευτικών δογμάτων, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να... Τι να σας πω τώρα, εδώ έχω ένα προβληματάκι ή μάλλον θα ήθελα μεγαλύτερη γλωσσική σαφήνεια. Δεν νομίζω ότι είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναμειχθεί στην ερμηνεία των ε, θρησκευτικών δογμάτων ε, που βεβαίως ε, ακριβώς λόγω του δογματισμού των δογμάτων που είναι βεβαίως κάτι προφανές δεν μπορούν να ερμηνευθούν πάρα πολύ εύκολα. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε οτιδήποτε κακή χρήση τέτοιου είδους αντιμετωπίσεων για πολιτικούς λόγους. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να είναι σαφέστερη η διατύπωση, κάποια γλωσσική καθαρότητα εδώ έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι ε, μπερδευόμαστε, ότι ε, υπάρχει οποτίποτε ανάμιξη ε, στην πολιτική ας πούμε διάσταση των θρησκειών. Να μην αφήσουμε κανένα ενδεχόμενο διαφορετικής ερμηνείας των θρησκευτικών δογματικών αρχών. Γιατί φοβούμε ότι μπορεί να υπάρξει δυνατότητα χειραγώγησης αυτών των ερμηνεών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στίερ. Μαριέτα, θέλεις να απαντήσεις, θέλεις να πεις κάτι, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι μια τροπολογία συμβιβαστική η οποία προήλθε από το αμυγές κείμενο, το δικό μου κείμενο και διάφορες τροπολογίες και έχει γίνει κάποιος συνδυασμός. Ε, τώρα αυτό το που αναφέρει ο κύριος συνάδελφος ε, το more open and inclusive interpretations of religious dogma in those countries and governments of which promote or condone and views of religion and culture εντάξει αυτό είναι μια γενικότερη τάση και επιθυμία που προέρχεται όμως από το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωσης θέλουμε να ασκείται με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και ανεξάρτητα από θρησκείες και θρησκευτικές πεπιθήσεις που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ελεύθερες αλλά δεν μπορεί να ασκείται μέσω αυτών ε, και επειδή γράφουμε σε άλλο σημείο ότι δεν πρέπει να θεωρούνται ως δικαιολογίε ε, οι θρησκευτικές και πολιτιστικές διαφορές για εξτρεμιστικές δραστηριότητες νομίζω ότι με αυτό πηγαίνει. Δεν βλέπω άλλο τρόπο ε, να συνδυάσουμε το καθαυτό κείμενο με, το, ε, με τις ε, τροπολογίες που υπάρχουν εδώ. Και δεν νομίζω ότι δημιουργεί κανένα πρόβλημα γιατί η έννοια δόγμα βέβαια οι θρησκείες και μάλιστα αυτές που η ερμηνεία τους χρησιμοποιείται για χειραγώγηση είναι δογματικές έχουν δογματικές αρχές και άκαμπτες αρχές. Είναι προφανές και όλες οι θρησκείες βέβαια έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, δογματικές αρχές και γι' αυτό ακριβώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα. Εγώ δεν βλέπω κάποιο τρόπο να πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Thank you very much, ε, ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα. Λοιπόν, η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας για αυτή την έκθεση προβλέπεται για αύριο το πρωί και αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, αυτό ήταν το τελευταίο θέμα μας στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Σας εύχομαι λοιπόν ε, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τελειώσαμε για σήμερα. Γεια σας.